Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην έκθεση της κυρίας Βέιμπερ για το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Βέιμπερ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέμε ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου αλλά μας αρέσει η κατάσταση την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν λόγοι που η κατάσταση διαμορφωθεί έτσι και που πρέπει να μας ανησυχούν. Σε, κάποια, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ την Επίτροπο Κρούς για την υποστήριξή της για το, στον πλουραλισμό και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο για όλους τους επιτρόπους. Αλλά δυστυχώς το, η έκθεση αυτή έγινε ακριβώς επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να δει έντονο ανώτερη αντίδραση από πλευράς Κομισιών και ιδιαίτερα από τον Επίτροπο των Αρμόδιων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το άρθρο 2 της συνθήκης και το άρθρο 11 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστηριχθούν από την Κομισιόν ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμη. Ελπίζω να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα οποία ζητούμε στην έκθεσή μας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη γιατί όχι μονάχα γιατί είμαστε εμείς οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών αλλά γιατί η έκθεση αυτή φτιάχτηκε μετά από πολλές μα πάρα πολλές ώρες διαβούλευση και σκέψεις. θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουν και να προωθήσουν μια δημοσιογραφία διερευνητική και ηθική οι δημοσιογράφοι είναι όλο και περισσότερο θύματα πίεσης, βίας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους δημοσιογράφους να μπορούν να εκφράζονται εύκολα. Επίθεση κατά δημοσιογράφου θα πρέπει να θεωρείται επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου και γι' αυτό θα πρέπει αμέσως να διαρευνάτε και να τιμωρείτε. Σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υπάρχει διαφανής και σταθερή νομοθεσία που θα προστατεύει τους δημοσιογράφους και τις αποστολές τους. Θα πρέπει να αποφύγουμε περιπτώσεις σαν και αυτές που βλέπουμε στη δική μου τη χώρα της Ρουμανίας όπου 7 χρόνια όπου εδώ και 7 χρόνια πολλά χρόνια που δεν τιμωρείται η δυσφήμιση έχουν γίνει τώρα προσπάθειες ε, να αλλάξει τα πράγματα και ε, γίνεται τώρα κουβέντα για την αποποινικοποίηση του αδικήματος αυτού της κοφαντίας και της δυσφήμισης. Είναι παράξενα αυτά που συμβαίνουν συμβαίνουν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε, ε, να είμαστε προσεκτικοί επίσης σχετικά με τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να απλώς να γράφουν καλά πράγματα για τους πολιτικούς ή για μας. Πρέπει να γράφουν την αλήθεια και πρέπει να τους βοηθούμε να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά λέμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Λούχαν για το 666. Για το 666. Μπορείτε να μετακινηθείτε αν θέλετε. Δεν τη διάλεξα εγώ τη θέση αυτή, με 666. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ την κυρία Βέμπερ για την έκθεσή της. Τη συγχαίρω για τη δουλειά που έκανε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται τα Ε είναι παρόμοια στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό αυτή η έκθεση για θέση προτύπων για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κίνητρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να είναι πιο θαραλέα στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά κανονισμούς για το θέμα αυτό. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τα εμπορικά ΜΜΕ. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στον αφορά τις πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα των δικαιούχων των ΜΜΕ. Αυτό θα ήταν υποφελές για τους πολίτες. Έτσι οι πολίτες μπορούν να διαθέτουν περισσότερες ε, πληροφορίες σχετικά με αυτά που προσφέρονται. Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στο μηχανισμό που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να εφαρμόζουν, λέει, τα κράτη-μέλη τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνει το πλουραλισμό των ΜΜΕ, η ίση πρόσβαση στις πληροφορίες και να δίνονται τα αναγκαία εχέγγυα για την ελευθεροτυπία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή και σαφής και σίγουρα αναφέρεται, αναφέρονται σε αυτήν ε, τη, στήριξη και, που, και, που μπορούμε να δώσουμε όλοι και εμείς και τα κράτη-μέλη και τα λοιπά. Ομόφωνα ψηφίστηκε η έκθεση στην Επιτροπή. Ε, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε τις βασικές μας αρχές και ελευθερίες και ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης είναι τα όργανα με τα οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ε, αξίες μας και τις αρχές μας. Γι' αυτό χρειάζεται ευρωπαϊκή υποστήριξη των δημοσιογράφων ε, και ε, και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, έγιναν πάρα πολλά θετικά σχόλια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Επίτροπο για το θέμα αυτό. Ε, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Βέμπερ, την εισηγήτρια. Είναι μια έκθεση που την περιμέναμε καιρό. Αρκεί να θυμηθείτε ότι η έκθεση αυτή έρχεται στην Ολομέλεια μετά από μακρές συζητήσει για την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία και στην Ουγγαρία. Βέβαια δεν περιοριζόμαστε, δεν, δείχνω το δάκτυλο μόνο αυτές τις δύο χώρες, διότι συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία. Γνωρίζουμε επίσης ότι η πραγματική δημοκρατία είναι εφικτή μόνο αν είναι ελεύθερος και ο τύπος. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βέβαια δεν είμαστε εδώ για να λέμε στους δημοσιογράφους τι πρέπει να κάνουν ή να μην κάνουν. Δεν υπαγορεύουμε εμείς τη διοντολογία, την ηθική τους, δεν είναι δικό μας, δική μας δουλειά. Δική μα δουλειά είναι να επαγρυπνούμε ώστε να έχουν την ελευθερία να γράφουν αυτά τα οποία επιθυμούν και να μπορούν οι πολίτες να επιλέγουν μεταξύ των διαφόρων εντύπων ή μέσων ενημέρωση και να υπάρχει πλουραλισμός. Το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση αυτή που ελπίζω να εγκριθεί αύριο με μεγάλη πλειοψηφία είναι ε, το εξή. Μπορούμε πλέον, αφού υπάρχει, θα εγκριθεί αυτή η έκθεση, ελπίζουμε με πλειοψηφία να έχουμε τα μέσα ώστε να το μεταφέρουμε στην νομοθεσία αυτό και να μπορούν πια να γράφουν οι δημοσιογράφοι αυτά που θέλουν να γράφουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιετρόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή, στο σημείο 31, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ελέγξει το πώς δίδονται οι άδειες στις εταιρείες που τους παρέχουν υπηρεσίες ε, διάφορες εκπομπές και κατά πόσο συμμορφώνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά την αδειοδότηση και κατά πόσο είναι ελεύθερα τα ΜΜΕ τα καθολικά στην Πολωνία. Εμποδίζονται οι δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου καναλιού του Γκρφάμ έστειλα στην Επίτροπο Κρούς ήδη μία επιστολή, με υποστήριξε και την ευχαριστώ, αλλά το τελευταίο εξάμεινο ε, δεν είδαμε αποτελέσματα. Πρόσφατα έγινε μια ειδική ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορούσε διακριτικές πρακτικές κατά των καθολικών ΜΜΕ στην Πολωνία. Οι πολιτικοί και οι πολίτες στην Πολωνία συνέλεξαν 2 εκατομμύρια υπογραφές κατά αυτών των διακρίσεων. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα εν πρώτης. Ευχαριστώ. Ο Ζήμπροφ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα της ελευθερίας των ΜΜΕ είναι θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χωρίς ελεύθερα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχουν πρότυπα ε, που αποτελούν και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δυστυχώς, πέρα από κάποια λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά το θέμα αυτό και γι' αυτό ανησυχούμε πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να κατανομάζουμε τις χώρες όπου απειλούνται τα μέσα ενημέρωσης και να κάνουμε όλο αυτό, αλλά πρέπει να παρεμβαίνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κάθε φορά παραβιάζεται η ελευθερία των ΜΜΕ ή που περιορίζεται. Θα πρέπει να πάρουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά. Είναι θεμελιώδης αρχή. Είναι βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελευθερία των ΜΜΕ. Ο καθηγητής Πιετρόφσκι που μίλησε πριν από μένα αναφέρθηκε στα προβλήματα με την αδειοδότηση των σταθμών, κάποιων τηλεοπτικών σταθμών στην Πολωνία. Και είναι πραγματικό πρόβλημα και δεν υπάρχει αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε τα ίδια πρότυπα να εφαρμόζονται σε όλου, κυρία Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βέιμπερ. Θα ήθελα να τονίσω ένα θέμα, το, ε, το θέμα της ε, ουδετερότητας των δικτύων που αναφέρεται στην έκθεση αυτή ε, ο όρος μία, φορά όμως και δεν τονίζεται ιδιαίτερα ε, γιατί τονίζω την, τον όρο αυτό ε, γιατί ε, ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή ότι όλα ψηφιοποιούνται όχι μόνο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ψηφιακοί αλλά τα βιβλία, η μουσική όλα αυτά ε, ψηφιοποιούνται αυτή τη στιγμή και γίνεται δηλαδή μια μετα τροπή αυτών των δημιουργημάτων γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ουδετερότητα σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Επίτροπε, κυρία Σαΐα, είπαμε ότι είναι θεματοφύλακα εξουσίας τα ΜΜΕ και η ανεξαρτησία των ΜΜΕ είναι χαρακτηριστικό σήμα της δημοκρατίας. Η ελευθερία λοιπόν των ΜΜΕ δεν πρέπει να απειλείται από περιορισμούς. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Η δημοκρατία προβλέπει ελευθερία έκφρασης και ο κόσμος μπορεί να έχει πληροφορίες και αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να τα απολαμβάνουν και τα σύγχρονα ΜΜΕ όπως και διάφοροι μηχανισμοί αναζήτηση στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα. Διάφοροι φορείς, τα κράτη-μέλη παρακολουθούν κατά πόσο υπάρχει αυτή η ελευθερία και ενημερώνουν σχετικά. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσπαθεί να εξασφαλίσει τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης πολύ συχνά εξετάζει το θέμα των ΜΜΕ. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι ένα από τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Κριτήρια που επιβάλλονται στις υποψήφιες χώρες που να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο teljes mértékben egyetértek weber jelentésével Συμφωνώ 100% με την έκθεση της κυρίας Βέιμπερ. Πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακαλέσει να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα εξασφαλίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Είμαι υπέρ επίσης της εποπτείας και των στα διάφορα κράτη-μέλη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ε, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Στην ε, Ουγγαρία ε, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Βεβαίω η κυρία Κρούς ξέρει ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές αλλά τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα της χώρας λένε ψέματα, ψεύδεται, ε, ψεύδονται οι δημόσιοι σταθμοί και δημόσια τηλεόραση στη χώρα μου. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Αξίζει τις υποστήριξής μας λέει Υπάρχουν και κάποια ε, σχόλια για τα δημόσια μέσα. Την ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η Επιτροπή ε, Πολιτισμού ε, και εγώ στηρίξαμε κάποιους παραγράφους στο κείμενο για τα δημόσια μέσα. Βελτίωση υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει αυτό την οικονομική κατάσταση. Υπάρχει ένα στελεοπτικό σταθμό στο Τερφάμ, το ανέφεραν συνάδελφοί μου πριν. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργό Μεταφορών ζήτησε εγγύηση 8 εκατομμυρίων ευρώ από μία εφημερίδα. Γιατί έγραψε για τα ρολόγια που φοράει, τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά από όσα παίρνει ως αμοιβή. Επίσης, ε, ε, ο Πρωθυπουργό μας προσέφυγε στα δικαστήρια κατά μίας ε, εφημερίδας για ένα σχόλιο, για ένα ανέκδοτο για την 1η Απριλιά. Και πάνε για αυτή την πλάκα ουσιαστικά την εφημερίδα στα δικαστήρια. Θέλω να ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και στρέφουμε προς την Κομισιόν. Παρακαλώ, κοιτάξτε τι γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες. Βλοβιέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από τρία χρόνια, κυρίες και κύριοι, εγκρίναμε την οδηγία για τις υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα. Είμαστε στο σωστό δρόμο, μεν, αλλά η συγγήτρια αναφέρει ότι δεν προστατεύονται παρκώς οι ανήλικοι υπάρχει επιβλαβές περιεχόμενο ε, στα μέσα ενημέρωσης ε, και τους επηρεάζει τους ε, ανηλίκους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερες ρυθμίσεις και θα πρέπει να υιοθετήσουμε, για να προστατεύσουμε τα παιδιά και να υιοθετήσουμε ήπια μέτρα, μη δεσμευτικά, για τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Παραδείγματο χάρη κάποιε τραδιαφημίσεις που ε, παραπλανούν ότι αυτή την περιεκτικότητά του ε, σε νάτριο ή σε ε, λιπαρά ή κάποιοι που διαφημίζουν προϊόντα ότι είναι για διαβητικούς ή δεν ξέρω γιατί, αλλά οι γιατροί λένε προσοχή γιατί μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή αυτά τα τρόφιμα. Πρόεδρος, μήπως θα σταματήσουμε να τρώμε και κρέας όπως έκανα εγώ. Θα ήταν μια καλή λύση για αυτή. Ο επόμενος είναι ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα της ελευθερίας του τύπου είναι πολύ σημαντικό θέμα, πολύ περίπλοκο, πολύ ευαίσθητο και διότι οι περιορισμοί σχετικοί παράγονται σε διαφορετικά επίπεδα και δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν κυρίω από μια επιφανειακή αναγνωσή τη κατάσταση. Υπάρχουν ελευθερίες που περιορίζονται μέσω νομοθετικών πράξεων Όπω έγινε στην Ουγγαρία. Υπάρχουν άλλε ελευθερίε που συνδέονται με διάφορε διαδικασίε συγκέντρωση και δίκε για συγκέντρωση που πλήττουν του πιο αδύναμους και του πιο μικρού. Και αυτά δεν τα γίνονται αμέσω αντιληπτά. Και μετά υπάρχουν ελευθερίε που προ... λόγω συγκρούσεων συμφερόντων ε, δημιουργούνται προβλήματα. Είναι κάποιος που χειρίζεται τα μέσα επικοινωνίας και διάφορους θεσμικούς φορείς και πολιτικούς φορείς. Έγινε επανειλημμένα αυτό τα τελευταία χρόνια στη χώρα μου. Ε, πιστεύω ότι όλες αυτές οι μορφές θα πρέπει να συνοδεύονται από αυξανόμενη προσοχή που θα δίνουμε όσον αφορά το δίκτυο. Πολλές επικοινωνίες περνούν από εκεί, από το διαδίκτυο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε διαδικασία που θα εγγυάται την πλήρη ελευθερία σε όλους και να μην περιοριζόμαστε μόνο στις παραδοσιακές μεθόδους διάδοσης των μέσων ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξυπακούεται ότι μία από τι θεμελιώδει αρχέ τη δημοκρατική κοινωνία είναι η ελευθεροτυπία. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω θέλουμε να έχουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Σε κάθε κράτο μέλο υπάρχουν διάφοροι τρόποι βέβαια για την εξασφάλιση ελευθεροτυπία και πώ την χειρίζονται την ελευθερία του τύπου. Ακούμε κάποιοι που έχουν τα μέσα να ελέγχουν το περιεχόμενο, οι εκδότες να ελέγχουν πάρα πολύ τους δημοσιογράφους και στον τύπο και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να συζητηθούν. Ε, υπάρχουν και ευθύνε που έρχονται με την ελευθερία όμως, κυρίως όσον αφορά την παρουσίαση των όσων συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια μήμοι με μεροληπτούν και αυτό το λιγότερο μπορώ να πω δεν είναι επαγγελματικά μέσα και παρουσιάζουν τα πράγματα πολύ αρνητικά. Χρειάζονται δίκαιες συνθήκες και ύψες προδιαγραφές και για την ελευθερία της έκφρασης και το πώς εφαρμόζεται η ελευθεροτυπία. Θα πρέπει να έχει τελικά και ο τύπος να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα σωστά για να έχει το κατάλληλο κύρος. Κυρία Τανσίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της Κοπενχάγης και εκεί συμπεριλαμβάνεται και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 11 εκεί λέγεται ότι πρέπει να διαφυλάσσεται η ελευθερία και ο πλουραλισμός των ΜΜΕ. Οι δημόσιες, ε, οι σταθμοί έχουν θεσμικό ε, θεσμική υποχρέωση να δίνουν στο κοινό πληροφορίε υψηλή ποιότητα, αξιόπιστε πληροφορίε, επαρκεί πληροφορίε και να είναι ανεξάρτητα τα μέσα αυτά, να μην επηρεάζονται πολιτικά συμφέροντα και εξωτερικέ πιέσει. Τα ιδιωτικά μέσα υπέχουν παρόμοιε υποχρεώσει όσον αφορά την ενημέρωση και τι πληροφορίε. Άρα πρέπει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα δίκαιο όπου τα ιδιωτικά μέσα και τα δημόσια μέσα να παίζουν το ρόλο που τους αρμόζει και να εγγυώνται την ανεξαρτησία όσον αφορά την παρουσίαση των ειδήσεων. Να μην δημιουργούνται μονοπόλια στον τομέα αυτό, στον τομέα των ειδήσεων και των διαφόρων υπηρεσιών που παρουσιάζουν τις ειδήσει και συγχαρητήρια στον εισηγητή για την έκθεση. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Η συνάδελφό μα, η κυρία Ρενάτε Βέμπερ, συνέταξε μια έξοχη έκθεση όσον αφορά τον πλουρισμό των μέσων και την ελευθερία των μέσων και είναι μια έκθεση που ταιριάζει στην όλη κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή συνθήκη Σαββόνα. Θα πρέπει επιτόπου να δούμε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν πλέον τα μικρά ΜΜΕ, δεν υπάρχουν τοπικά νέα. Όλα ενδιαφέρουν όλου του Ευρωπαίου πια. Ε, η διακυβέρνηση στην Ευρώπη ενδιαφέρει όλου. Είναι τεράστιο ο τομέα και θα πρέπει να συζητήσουμε την ελευθερία των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη, ώστε η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να λειτουργεί πραγματικά. Αυτό το σχόλιο ακούστηκε από την ομάδα υψηλού επίπεδου, τη οποία προεδρεύει η Επίτροπο κυρία Κρού. Έχουν δοθεί καινούρια κίνητα τι εργασίε αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία. Αυτό περιμένουν οι πολίτε. Νομοθεσία για τα ΜΜΕ. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τις επιφανειακές συζητήσεις περί επικουρικότητας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρόσβαση τι πληροφορίε, το δικαίωμα που έχουν οι δημοσιογράφοι να είναι ελεύθεροι. Και όλα αυτά θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ρενάτε Βέιμπερ για την έκθεσή της και ευχαριστώ και τους ε, βουλευτές πήραν μέρος στη συζήτηση που μόλις έγινε. Πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία την ψηφοφορία αύριο και πραγματικά φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα μας δώσει προοπτικές για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της ελευθεροτυπίας και του πλουραλισμού στην Ευρώπη και είδαμε την περασμένη εβδομάδα λόγω χάρη στις Ηνωμένε Πολιτείε ότι και εκεί υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις ε, σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφικής ελευθερίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε απειλή στην ελευθεροτυπία εδώ στο Κοινοβούλιο πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι η ελευθεροτυπία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας μας και το θέμα έχει τεθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ε, δεν είναι σωστό ο, Αλλά είναι γεγονός ότι δεν αρκεί να λέμε ωραία λόγια, πρέπει να παρέμβουμε. Αλλά για να παρέμβουμε πρέπει να έχουμε και τα μέσα και τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Χαίρομαι που αυτή τη φορά έχουμε εδώ μια σαφή έκθεση πολύ συγκεκριμένη η οποία άμα μας άμα υπερψηφιστεί θα, θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και με τα κράτη-μέλη να συζητήσουμε τι μπορούν να κάνουν και ποιοι πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για να διευκρινιστούν οι, Ευρω... οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο αυτές τις αρμοδιότητες. Και τρίτο και βασικό πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς χωρών μερών για να προχωρήσουμε. Χαίρομαι που ε, φαίνεται να υπάρχει ε, η βούληση από πλευράς της ε, τρέχουσας προεδρίας και η Λιθουανική Προεδρία ε, θα ασχοληθεί με το θέμα τη σχετική ομάδα με υπό την προεδρία του τέος πρόεδρου της Λετωνίας ήδη συζήτησε θέματα πολλά σχετικά με την ελευθεροτυπία και, την, ε, ε, και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης και τελικά ε, κατέληξε σε 30 συστάσεις που μερικές από τις οποίες είναι παρόμοια με αυτά που λέει η κυρία Βέμπερ στην έκθεσή της. Πραγματικά θα πρέπει ε, να φροντίσουμε αυτά που προτείνονται και στην έκθεση Βέμπερ αλλά και στην έκθεση της, στα πορίσματα της ανεξάρτητης αυτής ομάδας υψηλού επίπεδου πρέπει πολλά από αυτά να τα εφαρμόσουμε πρέπει να υπάρχει ένας ειδικό προϋπολογισμός για την εφαρμογή τέτοιου είδους μέτρων θα μας δώσει τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να κάνουμε πολύ πιο σοβαρή δουλειά και θα πρέπει ίσως να δούμε και το θέμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ελευθερία του, των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός τώρα ο, που, σε λίγο και δύο δημόσιες διαβουλεύσεις έχουν ξεκινήσει επίσης πρόσφατα. Πρώτα-πρώτα για να δούμε, να συζητηθούν οι συστάσεις της ανεξάρτητης αυτής ομάδας υψηλού επίπεδου και δεύτερον για να συλλέξουμε τις γνώμες των ανεξαρτήτων αρχών που είναι υπεύθυνες για τα, ε, τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Ε, να δούμε ενδεχόμενη αναθεώρηση του άρθρου 30 του AMSD και η έκθεση της Ρενάτε Βέιμπερ πραγματικά φτάνει την κατάλληλη στιγμή είναι η σωστή χρονική στιγμή ε, αυτή για την έκθεση κυρίας Βέμπερ που ελπίζουμε να υπερψηφιστεί αύριο. Ο Άρα στο άμεσο μέλλον θα ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε και εκτός από και ελπίζω πρόεδρε να έχουμε και σαφή και συγκεκριμένα αποτελέσματα όπως θέλει και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο και τους συνεργάτες της. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους, ευχαριστώ την κυρία Βέμπρη για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, ρωτάει ο Πρόεδρος. Thank you all very much indeed. That debate is closed. The vote is Κλείνει η συζήτηση αυτή, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο 12 και μισή. Επόμενο θέμα η έκθεση του κυρίου Μπόρις για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.